των καταναλωτών. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέπχαρτ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι, αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην σε διάταξη είναι η σύσταση του κυρίου Λένε ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρασιτεχνίας. Τον λόγο έχει ο εισηγητής μας, ο κύριος Λένε, για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εδώ το θέμα είναι για δεύτερη φορά η ενισχυμένη συνεργασία. Τα στα θέματα οικογενειακού δικαίου. Πριν από κάποιους μήνες αποφασίσαμε σύμφωνα με τη, Λισαβόνα, με τη της Λισαβόνα στα θέματα ενισχυμένης συνεργασίας. Τώρα είναι δεύτερη φορά αυτή λοιπόν. Είναι θέμα διαδικαστικό και καθαρά μόνο διαδικαστικό. Το λέω αυτό και το τονίζω, δεν συζητάμε επί του περιεχομένου. Αυτό θα το συζητήσουμε σε μετέπειτα χρονική στιγμή. Να παρατηρήσω επίσης το εξής. Με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι η Ουγγρική Προεδρία σήμερα είναι εδώ. Είναι πρώτη φορά, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Προεδρία έρχεται Δευτέρα απόγευμα. Αυτό καταδεικνύει και τη σημασία του φακέλου αυτού. Από το 2001 συζητάμε τέτοια θέματα ευρωπαϊκών ευρεσιτεχνιών βάσει μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο νομίζω με μια έκθεση τοποθετήθηκε με σαφήνεια σε ό,τι αφορά την πρώτη ανάγνωση. Και δεν ήταν εύκολο όμω να βρεθεί συμφωνία στο Συμβούλιο. Δύο προβλήματα είχαμε. Καταρχά, θέματα δικαιοδοσία, ε, ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο, αλλά και το θέμα τη γλώσσα. Το θέμα της δικαιοδοσίας μπορεί να επιληθεί σύντομα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί θα ληφθεί αρχές Μαρτίου και τελικά θα καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε προχωρήσει όμως στο θέμα των γλωσσών. Η Βελγική Προεδρία διαπίστωσε το φθινόπωρο πέρσι ότι ε, σε ό,τι αφορά τη γλωσσική διαμάχη δεν ήταν δυνατόν να βρει μια λύση τουλάχιστον όχι στα πλαίσια της ομοφωνίας που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας γιατί είναι εκ διαμέτρου διαφορετικές οι απόψεις μεταξύ των αρχών, για παράδειγμα ότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 23 γλώσσες με ίδια δικαιώματα και του γεγονότος ότι ε, μία, μία δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και μετάφραση σε όλες τις γλώσσες συνεπάγεται τεράστιο κόστος. Άρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ε, πέρα από το θέμα της ε, νομικής ισχύως της μετάφρασης, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με το σύστημα αυτό γιατί είναι υπερβολικά ακριβό σε ό,τι αφορά τη μετάφραση. Γιατί μια τέτοια ευρεσιτεχνία με πολλέ γλώσσε είναι ένα θέμα που μπορούν νομίζω να αντιμετωπίσουν μόνο οι μεγάλε επιχειρήσει στα μεγάλα κρατημέλη και όχι οι μικρέ επιχειρήσει. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλέ φορέ σε ψηφίσματα είχε προετοιμάσει κάποιες πρόοδους, είχε ζητήσει πρόοδους. Νομίζω ότι τώρα πια όμως έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Η ε, Προεδρία ζήτησε από την Κομισιόν να προετοιμάσει μία πρόταση σχετική. Η Κομισιόν ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή. Το Συμβούλιο μας ζήτησε την ε, γνωμοδότησή μας. 16 προς 5 ε, ψήφους ψήφισε η Αρμόδια Επιτροπή. 25 κράτη-μέλη στηρίζουν την πρόταση αυτή τώρα πια και θα έλεγα ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να κάνουμε ένα βήμα προ τα προς και το Κοινοβούλιο να δώσει την ε, σύμφωνη γνώμη του για τη διαδικασία αυτή για να δούμε επιτέλου το φω στην έξοδο του τούνελ. Και θα τελειώνω λέγοντα τα εξή. Δεν έχουμε πολλού πόρου φυσικού στην Ευρώπη. Αυτό που έχουμε είναι ο εγκέφαλός μας, η δημιουργικότητά μας, οι ιδέες μας και αυτέ θα πρέπει να τις προφυλάξουμε. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε έναντι της Κίνας, της Ινδίας και άλλων αναπτυσσομένων μεγάλων χωρών στον κόσμο να πούμε ότι θα πρέπει να προστατεύεται την πνευματική ιδιοκτησία που μπορούμε να το κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς μια ε, ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία και γι' αυτό κάνω έκκληση να υποστηρίξετε αυτή την πρόταση για μια ενδυναμωμένη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας εξ του Συμβουλίου, η κυρία Γιώρη. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, είναι ένα κακό θέμα. Λοιπόν, ε, είναι μεγάλη τιμή για μένα που απευθύνομαι στους βουλευτές σήμερα. Όπως μόλις μας είπε ο κύριος Λένε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και άρα είναι εξίσου σοβαρή και η στάση του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την επικοδομητική του στάση. Στήριξε το Συμβούλιο στι προσπάθειε που κάνει ώστε να υπάρχει επαρκή προστασία με διπλώματα ευρεσιτεχνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προωθούμε λοιπόν την συγκρότηση ενό ενιαίου συστήματο έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Δεύτερον, σήμερα το πρωί το Συμβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε να ζητήσει την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δρομολογηθεί ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό. Εάν δώσετε τη σύμφωνη γνώμη στι 10 Μαρτίου, το Συμβούλιο Ανταγωνισμού ε, θα δώσει την έγκριση και θα, ε, την σχετική άδεια για να δρομολογηθεί η διαδικασία. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ένωσης. Φέρουμε την ευθύνη διότι η καινοτομία είναι βασική κινητήριος δύναμη της ανταγωνιστικότητας όχι μόνο στην Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξ αρχής ήταν σαφές ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που εξυπηρετούν αυτό το στόχο είναι η δημιουργία ενό ευρωπαϊκού διπλώματο ευρεσιτεχνία. Έχει σημειωθεί βέβαια καθυστέρηση άνω των 30 ετών. Ε, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την καθεστική ατάξη. Εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για τι μεταφράσει και για τι διοικητικέ διαδικασίε για να κατοχυρώσει κάποιο προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνία στα 27 διαφορετικά νομικά συστήματα. Ενώ στη ΣΥΠΑ ένα εφευρέτη μπορεί για όλη την Αμερικανική επικράτεια να αποκτήσει δίπλωμα ε, για 1.850 ευρώ συνολικά στην Ένωση. Το αντίστοιχο ποσό είναι 20.000 και ισχύει στην επικράτεια 13 μόνο μελών της Ένωσης. Βάσει των υπολογισμών που έχουμε κάνει, ε, ε, 7 με 8 εκατομμύρια ε, ευρώ ε, χάνονται από τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω αυτής της κατάστασης και φυσικά μπορεί να σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στην τεχνολογική κυρίως πρόοδο να κατοχυρώσουμε ένα ενιαίο δίπλωμα. Δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοια προστασία. Δηλαδή, ο όποιος υποβάλλει αίτηση αντιμετωπίζει 27 διαφορετικές ένομες τάξεις. Οπότε η προστασία ισχύει συνήθως σε ένα μόνο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών που προστατεύονται από τα διπλώματα στην επικράτεια κάποιων κροτών ενώ σε άλλα όχι. Σαφώς προτιμούσαμε ανέκαθεν ένα πραγματικό δίπλο, ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα ισχύει στην επικράτεια των 27 κρατών μελών. Λυπούμεθα βαθύτατα για την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς και τις μεταφράσεις. Ε, δεν ε, απέδωσαν καρπούς και δεν καταλήξαμε, δεν θα, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον δεν θα καταλήξουμε σε συνενετική λύση για αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω επίσης ότι οι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται ε, σοβαρή πίεση για να σημειωθεί πρόοδο, ε, γιατί έχουμε τον πίνακα βαλογία που εσχάτω δημοσιεύθηκε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δείχνει τα κενά που έχουμε σε σχέση με την Ιαπωνία, παραδείγματο χάρη για την καινοτομία και τι νέε τεχνολογίε. Και οι αναδυόμενε οικονομίε έχουν φτάσει σχεδόν στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνία έχει προφανή σημασία πέρα από αυτό το ζήτημα και έχουμε αυτό το το κατακαιρματισμένο σύστημα που φυσικά δεν θέλει ε, τους αλλοδαπούς και δεν είναι ανταγωνιστικό. Στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών θεωρεί ότι η δημιουργία μια ενιαία προστασία, στα πλαίσια τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία είναι μονόδρομο προ το παρόν. 27 κράτη-μέλη έχουν υποβάλει σχετική αίτηση ούτω ώστε να κινηθεί η διαδικασία της ενισχυμένης διαδικασίας ε, και αναμένουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να έχουμε κάποια ικανοποίηση ικανοποιητικά αποτελέσματα ε, και ε, καταβάλλονται κάθε προσπάθειες από την Επίτροπο για να ε, σημειωθεί πρόοδος. Υπάρχουν βέβαια ενστάσεις και αμφιβολίες κυρίως από την Ισπανία και από την Ιταλία και θα ήθελα να στραφώ στους Ισπανούς και Ιταλούς βουλευτές στη μητρική τους γλώσσα. Καταρχήν, Προς τους Ισπανούς βολευτές πρέπει να πω ότι μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας και με τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος προστασίας των διπλωμάτων θα προχωρήσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Και τώρα προς τους Ιταλούς φίλους μας. Όπως και να έχει το πράγμα, θέλω να υπογραμμίσω για να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση. Καμία επιχείρηση και κανένα άτομο, άσχετα από το κράτος προέλευσης, θα αποκλείεται από τα ευεργετήματα του μελλοντικού διπλώματος, ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω και να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η έγκριση που προτείνει ο κύριος Λένε για, το, για την ενισχυμένη συνεργασία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, τους Ευρωπαίους εφευρέτες να τους βοηθήσουμε με μια ενιαία πλέον προστασία των ευρυσιτεχνιών τους στην Ευρώπη. Είναι κάτι το απαράβατο για τον ανταγωνισμό στην Ήπειρό μας και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει γι' αυτόν τον λόγο εμείς να προστατεύσουμε τις εφευρέσεις, τις δημιουργίες κυρίως στον βιομηχανικό τομέα. Στις 13 ε, ε, Ιανουαρίου του 2010 αλλά και άλλες φορές δεσμεύθηκα να προωθήσω αυτό το ντοσιέ για να εκπληρώσω και τις επιθυμίες του προηγουμένου, του προκατόχου μου επιτρόπου. Με την συνεισφορά της Βελγικής Προεδρίας βελτιώσαμε το σχέδιο. Δεν πετύχαμε βέβαια την ομοφωνία όπως θα θέλαμε για αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν, στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας είπαμε να θεσπίσουμε το καθεστώς ενισχυμένης συνεργασίας. 12 κράτη-μέλη αρχικά, όπως είπε και ο κύριος Λένε, είχαν προτείνει την ενισχυμένη συνεργασία και σήμερα είναι 25 που την προσυπογράφουν. Η Ουγγρική Προεδρία μετά την Βελγική επέδειξε ιδιαίτερη βούληση στο να ολοκληρώνουμε με αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Λένε και την Επιτροπή σας, την Νομική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για το ρόλο που παίξατε όλοι για να προωθήσουμε αυτό το ντοσέ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Κομισιόν θέλει στην ενισχυμένη συνεργασία να εισχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη. Εγώ ελπίζω ότι τελικά όλα τα κράτη θα υποστηρίξουν αυτή την πρόταση η οποία είναι πολιτικά αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη αλλά και οικονομικά απαραίτητη από όλες τις επιχειρήσεις. Και αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους εφευρέτες. Εγώ ως αρμόδιος επίτροπος θα περιφρουρήσω ούτω ώστε να παραμείνει η ενισχυμένη συνεργασία συμβατή με τις συνθήκες και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όπως πολύ σωστά η υπουργό είπε στα Ισπανικά και στα Ιταλικά, αυτή η προστασία λοιπόν μέσω των, ε, των, ε, της, της Ευρωπαϊκής Ευρυσιτεχνίας θα προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη και τα πλεονεκτήματα θα είναι τα ίδια για όλους τους εφευρέτες και για όλες τις ε, καινοτόμες επιχειρήσεις της Ένωσης διότι και το κόστος θα ορθολογικοποιηθεί αλλά και το κόστος της μετάφρασης θα μειωθεί. Εμείς ε, αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις οικονομικές επιπτώσεις του μέτρου. Δυστυχώς δεν πετύχαμε ακόμα να έχουμε συμφωνία των 27, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η ενισχυμένη συνεργασία. Και αυτό όταν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο για να αποφασίσει και τα τελευταία μέτρα για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με αυτή τη νέα προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προκαταβολικά για την υποστήριξη αυτού του σχεδίου. Σας ευχαριστώ Επίτροπε κυρία Μπέρνια. Επόμενη οι ομιλητέ εξ των πολιτικών ομάδων, καρχική ο συνάδελφο Παλτασάνη για το κόμμα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Με έναν ιδιαίτερο δυναμισμό και ταχύτητα το Κοινοβούλιο θα δώσει το πράσινο φως για ε, την ενισχυμένη συνεργασία που αφορά στην εσωτερική αγορά. Το επιχείρημα είναι ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή ευρυσιτεχνία συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όμως μόνο στις 30 Ιουνίου του 2010 αποφασίστηκε το καθεστώς μετάφρασης και μόνο τότε το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ομοφωνία. Το ότι δεν υπήρχε και δυνατότητα ομοφωνίας σε ένα εγγυσμένος ρυθμοί του Κοινοβουλίου. Ελπίζω βέβαια να αποτελέσουν παράδειγμα και για το μέλλον, διότι καταρρίψαμε ρεκόρ για τη γρήγορη νομοθετική διαδικασία. Εμένα δεν είναι πρόθεσή μου να εκπροσωπήσω εδώ μόνο τη χώρα μου, που δεν συμφωνεί με την ενισχυμένη συνεργασία. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες αυτό το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρυσιτεχνίας για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Και θέλω να πω το στο σώμα για τη μελλοντική λειτουργία του συστήματος. Η ψήφος με, με το σύστημα της ενισχυμένης συνεργασίας θα θεσμοθετεί έναν τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς που θα έπρεπε κανονικά να είναι η τελευταία προσφυγή για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει στο μέλλον να εκφράζεται αυτό όνομα και εξαντλητικά και θα έπρεπε όλα τα μέτρα να είναι υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ των εφευρετών και όχι υπέρ του συμφέροντος ορισμένων χωρών. Ευχαριστώ κύριε Ζραπ και δύο λεπτά εξ ομάδα του. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, η αιτηλόγηση που έδωσε ο εισηγητής είναι σωστή. Δεν χρειάζεται να προσθέσει κανένα τίποτα και γι' αυτό και η ομάδα μου θα υπερψηφίσει την ενδυναμωμένη συνεργασία. Σε όλες τις πολιτικές ομάδες υπάρχουν κάποιες αποκλίνουσες απόψεις, νόμιμο, καλό να ακουστούν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο συγχητής, αυτό που είπε η Προεδρία του Συμβουλίου και αυτό που είπε και ο Επίτροπος, καταδεικνύουν ότι πραγματικά έχει φτάσει πια το πλήρωμα του χρόνου. Δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε άλλο. Δεν είναι αυτό που λένε ορισμένοι ότι βιαστήκαμε, χωρίς συζήτηση θέλουμε να προχωρήσουμε. Όχι. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι σωστό. Δεν συζήτησαμε το θέμα της γλώσσας από τότε που η Κομισιόν υπέβαλε την τελευταία της πρόταση πέρσι. Το θέμα των γλωσσών συζητιέται καμιά δεκαετία, αν όχι περισσότερο. Δεν είναι τίποτα το καινούριο και αν κανένας κοιτάξει τι ε, διαφορετικά μοντέλα προτάθηκαν τους τελευταίους μήνες και συζητήθηκαν δεν μπορεί πραγματικά να πει ότι δεν υπήρχε επακή συζήτηση. Πρέπει να προχωρήσουμε. Το δεύτερο επιχείρημα είναι καταστρέφουμε την εσωτερική αγορά. Μα στι ευρεσιτεχνίε δεν έχουμε εσωτερική αγορά. Πώς θα καταστρέψουμε λοιπόν κάτι που δεν υπάρχει. Και αν ξέρουμε, όπως ξέρουμε, ότι για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρειαζόμαστε ενιαία διπλώματα ευρυσεχνίας, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε στο status quo. Αλλά νομίζω θα προχωρήσουμε. Και το τρίτο επιχείρημα που ακούγεται συγκεκριμένα είναι ότι το Κοινοβούλιο, εάν συμφωνήσει με την ε, δαμωμένη συνεργασία, εγκαταλείπει αρμοδιότητες. Δεν είναι άλλη θέση αυτό. Για διαβάστε τη συνθήκη της Λισαβόνες για διαβάστε τον εσωτερικό μας κανονισμό. Δεν χάνουμε κανένα δικαίωμα, καμία αρμοδιότητα αν συμφωνήσουμε τώρα με την ενδυναμωμένη συνεργασία. Διατηρούμε όλα μας τα δικαιώματα. Διαβούλευση βέβαια όσον αφορά τις γλώσσες, γιατί αυτό είναι ομόφωνο. Συναπόθεση όσον αφορά τον κανονισμό για τις ευρεσιτεχνίες και σύμφωνη γνώμη όσον αφορά τις πατέντες πάλι. Λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτα του αντίον. Πρόεδρο, ευχαριστώ συνάδελφε Ραπκά. Επόμενο για δύο λεπτά, εξ ομάδα η κυρία Βίξτραμ. Ευχαριστώ. Αρχίζοντα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε. Εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο στον τομέα αυτό ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Μπαρνιέ γιατί ε, προώθησε το θέμα. Όπως ακούσαμε έχει συζητηθεί το θέμα επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες και τώρα είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να καταλήξει σε ομοθυμία που απαιτείται από συνθήκη από πλευρά του Συμβουλίου για να βρεθεί μια λύση. Πολλά κράτη-μέλη λοιπόν ζήτησαν να δρομολογηθεί ενισχυμένη συνεργασία ε, και θεωρώ ότι ε, προσκαλούμε όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στη διαδικασία ή αν το επιθυμούν βάσει της ενισχυμένης διαδικασίας. Οπότε το θέμα που τίθεται ε, σήμερα είναι το εξή. Θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη το Κοινοβούλιο σε αυτό το αίτημα του Συμβουλίου ή όχι. οι φιλελεύθεροι και εγώ προσωπικά πιστεύουμε ότι προφανώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του βάσει και των εισηγήσεων του κυρίου Λένε ε, ούτως ώστε ε, να προστατευθούν οι εφευρέσεις ε, για να προωθηθεί η καινοτομία, για να δημιουργηθούν νέα προϊόντα με τις νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να τονωθεί έτσι περαιτέρω η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης σήμερα. Για μια μικρή επιχείρηση ή για έναν εφευρέτη, έναν ιδιότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, χρονοβόρα για να καταχειρώσει την εφεύρεση του. Είπαμε στη ΣΥΠΑ, κοστίζει 1.800 περίπου ευρώ το δίπλωμα ευρεσιτεχνή, 11 φορέ παραπάνω κοστίζει στην Ένωση και σχεδόν 20.000. Πολυεθνικέ εταιρείε ε, με μεγάλου πόρου και νομική τεχνογνωσία προφανώ θα τα καταφέρνουν πάντοτε, όποιο και αν είναι το σύστημα. Ε, αλλά οι ιδιώτε, οι εφευρέτε, αυτοί πληρώνουν τα σπασμένα λόγω του σημερινού συστήματο. Οπότε ήρθε η ώρα, εν πάση περιπτώσει, να του προστατεύσουμε, γιατί ε, εκείνοι θα γίνουν οι μεγάλοι εργοδότε ε, του μέλλοντο. Ε, τους. χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε η ώρα, δεν έχουμε πια χρόνο για χάσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Βίξτρο. Δύο λεπτά εξ των Πρασίνων. Η κυρία Λίχτενμπεργκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνία κατά πάσα πιθανότητα σε ορισμένου τομεί τη οικονομία και τη επιστήμη θα είναι βελτίωση, παρόλο που πρέπει να πω ότι οι ελπίδες είναι κάπως υπερβολικές. Οι ελπίδες που τρέφει κανένας για αυτή την ευαισθηχνία. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε νομίζω. Εγώ θα μιλήσω εδώ κατά της ενισχυμένης συνεργασίας. Πρόσφατα είχαμε την υπόθεση με τα διαζύγια στην ενισχυμένη συνεργασία. Μετά από την απόφαση αυτή έχουμε το επόμενο θέμα στην ισχυμένη ε, συνεργασία. Εάν δώσουμε την έγκριση αυτή εδώ, έως όχι, θα δούμε να πολλαπλασιάζονται οι ισχυμένες ε, συνεργασίες, γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολη η οδός Επίτευξη συνένεση στο Συμβούλιο. Δεν ήταν αυτό που είχαμε κατά νου στην κοινοβουλευτική ε, συνέλευση όταν συζητήσαμε το θέμα της ενισχυμένης ε, συνεργασίας. Η καλύτερη κυβέρνηση που πολλοί τη συζητάνε έχει ένα στοιχείο που λέει διαφάνεια και σαφήνεια. Αυτά ε, εγκαταλείπονται μέσα στα πλαίσια της ενισχυμένης διαδικασίας, ε, συνεργασίας. Συγγνώμη. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι τεράστιο πρόβλημα για το μέλλον. Όταν έχουμε τα διάφορα θέματα που, για τα οποία έχουμε κάποιες υποομάδες κρατών που μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτά. Καλό να λέμε, έχουμε καλέσει και τους άλλους να συνεργαστούν, ναι, αλλά υπό ποιους όρους. Εγώ θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτή τη φορά Εν αντιθέσει με αυτά που έγιναν στο παρελθόν, θα υπήρχε ευκαιρία συμφωνίας εάν οι διαπραγματεύσεις είχαν διαρκέσει λίγο περισσότερο. Θεωρώ ότι η οδός της ενισχυμένη συνεργασίας στον τομέα των ευρεσιτεχνών δεν είναι σωστή άγουσα και γι' αυτό δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με την πρόταση που υποβάλλεται. Πρόεδρε, ευχαριστώ στην άλλη φίλη Ένα λεπτό εξ στη ΕΚΑΕΡ συνάδελφο Ευχαριστώ. Εδώ και χρόνια στην Ευρώπη Γίνεται μία συζήτηση για τα διπλώματα τεχνίας και οι επιχειρηματίες κρίνουν πως θα μειωθεί ε, το κόστος έκδοσης των διπλωμάτων στην επικράτεια της Ένωσης ε, με, αν εγκριθεί νέο σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, Αυτή την κατεύθυνση προκρίνει και ο εισηγητής μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με όλα τα αυτά ε, οφείλουμε να εξετάσουμε κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα της πρότασης. Ήδη ακούστηκε σήμερα το θέμα των μεταφράσεων, των μεταφράσεων των διπλωμάτων από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Θα γίνονται εφ' οι μεταφράσεις σε τρεις μόνο γλώσσες. Αυτό οφείλουμε να το επανεξετάσουμε. Γιατί σε τρεις γλώσσες και όχι σε περισσότερες. Ε, έτσι θα, οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν μόνο τις τρεις γλώσσες θα είναι πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστούμε. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε ήδη να δημιουργήσει ε, ένα Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ενδυστησίας όπου απορρίφθηκε ε, το, από το Συμβούλιο. Τώρα η Κομισιόν το Και αυτό είναι πάλι ένα παράδειγμα ε, μιας αυτοκρατορικής τάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό θα επιβερύνει ιδιαίτερα τις κοινοτομικές ε, επιθυμίες. Το θέμα προωθείται από 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν πλήττει κανένας ότι η Βρετανική κυβέρνηση προωθεί την πρόταση αυτή. Το κάνανε πάντα οι κυβερνήσει τη Μεγάλη Βρετανία αυτό, παρόλο που έδιναν εντύπωση ότι κάνουν το αντίθετο. Ευχαριστώ, συνάδελφε Πέτεν. Η υπόλοιπη ομιλητέ τώρα. Η συνάδελφο Γκάλο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από τη γένεσή της αναρωτιέται η ανθρωπότητα για τη ζωή και το θάνατο. Τώρα, από το 70 και μετά να μην έχει ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της ευρωπαϊκής έβριση τεχνίας ε, πραγματικά είναι απελπισία. Και πραγματικά χαιρετίζω εγώ τον ε, κύριο, τον κύριο Λένε για την προσπάθειά του και για την προσοχή που επέδειξε προς τους Ιταλούς και Ισπανούς συναδέλφους. Εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Σήμερα εμείς δεν πρέπει να αποφασίσουμε εδώ ένα γλωσσικό θέμα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Ιουλίου του 2010 επαφίεται στο γλωσσικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρυσιτεχνιών που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Αλλά όμως αυτή η γλωσσική συζήτηση δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Σήμερα μιλάμε οι 25 χώρες οι οποίες το θέλουν να προχωρήσουν μέσα από το σύστημα της ενισχυμένης συνεργασίας ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που πληρώνουν τις ευρυσιτεχνίες τους 11 φορές πιο ακριβά από ό,τι αμερικάνικες επιχειρήσεις. Πρέπει να επιδείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα είναι όριμο και ξεπέρασε τις μικροδιαμάχες πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση που μας περιμένει. Ας, σταματήσουμε πια να προχωράμε σημειωτών. Ας προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτήν την μεγάλη πορεία προς την ευρωπαϊκή Ευρωστηχνία. Ευχαριστώ συνάδελφο Γκάλα. Η κυρία Φλεξίδα Βαβένοβα δεν είναι παρούσα. Οπότε για ένα λεπτό ο συνάδελφος Κοτσούσνικ. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι βουλευτέ, ε, κύριε Πρόεδρο, ο κύριος Ομπάμα ε, στην ε, ετήσια ομιλία του τόνισε πόσο σημαντική είναι η καινοτομία στη ΣΥΠΑ και χαρακτήρισε ω Πούτνικ την καινοτομία στι μέρε μα και περνώντα έτσι ένα σαφέ μήνυμα τη σημασία που έχει, τη βαρύτητα που έχει η καινοτομία τόσο ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστική τη ε, θέση σε παγκόσμια κλίμακα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από τα βασικότερα εργαλεία τη καινοτομία για να υπερβούμε του τίγρε τη καινοτομία, ε, παραδείγματο χάρη την Κίνα και τη Βραζιλία, είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνία γιατί θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων χάρη σε αυτά και ω εκ τούτου είναι κέρια σημασία σε αυτό το εργαλείο αν θέλουμε να προωθήσουμε την ε, καινοτομία στην Ένωση. Ε, και υπάρχουν υποδέστερα θέματα όπως παραδείγματος χάρη προστασία των γλωσσών ε, και αυτό αποτελεί φραγμό για κάποια κράτη-μέλη. Ωραία, κάποια κράτη-μέλη δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. μην χάσουμε το Sputnik. Ε, τώρα ο κύριος White για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό όλων των γλωσσών βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι σεβόμαστε αυτές τις αρχές. Εμείς θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ευρυστεχνιών και συγχαίρω τον συνάδελφο λένε γι' αυτό και θέλουμε να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Τώρα, για ένα θέμα τόσο σημαντικό επιλέχθηκε από τη συνθήκη η ενισχυμένη συνεργασία που πρέπει να αποτελεί μόνο τελευταία δικλίδα. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ αντιβαίνουμε τα άρθρα 118 και 126 της συνθήκης ε, και έχουν αλλάξει οι όροι πλέον από ό,τι φαίνεται στο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε εμείς την ενισχυμένη συνεργασία να τη χρησιμοποιούμε για την Ευρώπη των διαφόρων ταχυτήτων. Ορισμένες χώρες που επιλέγουν αυτό το σύστημα θα υποστούν τις επιπτώσεις αργότερα. Και στο τέλος θα χάσουμε όλοι. Σας παρακαλώ λίγο πιο αργά. Πιο αργά παρακαλώ. <laughs> Το, τα ισπανικά τα μιλάνε 850 εκατομμύρια άνθρωποι. Από τις γλώσσες που προτείνεται για την ευρυσιτεχνία, μόνο μία είναι συγκρίσιμη με τα ισπανικά. Λοιπόν, 1850 ευρώ. Ε, ας αφήσουμε τότε μόνο τα αγγλικά. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το ευκαιριακό εδώ, συγκυριακό καθαρά. Είναι ένα πολιτικό κριτήριο πίσω, που κρύβεται πίσω από όλα αυτά και που συνδέεται με γραφειοκρατικά τερτύπια τα οποία θα επιβαρύνουν πολίτες και ισπανικές επιχειρήσεις. Όλα αυτά αντιβαίνουν με το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζονται στη γλώσσα τους. Πρόκειται λοιπόν για στρέβλωση του ανταγωνισμού, κατακαιρμάτιση της αγοράς. Πρόκειται για ατυπία, πρόκειται για μια παρανομία την οποία θα λύσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη όλες αυτές οι προειδοποίησεις. Γιατί δεν λύνεται η κατάσταση, δεν διορθώνεται προσφεύγοντας αυτό το οποίο λένε οι συνθήκες όπως ζητάει η Ισπανία. Σας ευχαριστώ Ζούρις Βάιτ. ένα λεπτό. Είναι απαράδεκτο Κύριε Πρόεδρε, να μην έχουμε μια ευρωπαϊκή ευρυσιτεχνία. Επιβαρύνονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δέκα φορές παραπάνω στοιχίζει η ευρυσιτεχνία στην Ευρώπη από ό,τι στη Ιαπωνία ή στην Αμερική. Επίσης και το copyright επί των ευρυσιτεχνιών έχει να κάνει με την, οικονομική, με την καθυστέρηση της οικονομικής ανάκαμψης. Και εμάς όμως δεν μας αρέσει το γλωσσικό καθεστώς. Αλλάζει όμως ε, το πολιτικό πλαίσιο γιατί 25 από τις 27 χώρες προσχωρούν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία προσπάθεια βοηθώντας και τα Ιταλικά, αξιολογώντας και τα Ιταλικά. Θέλουμε να προστατευθεί η Ιταλική γλώσσα. Αλλά η κυβέρνησή μας έχει κόψει τα κονδύλια σε αυτόν τον τομέα. Και σίγουρα θα το παλέψουμε. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Συνάδελφος μα είπε Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή η διαδικασία είναι ένα μοντάζ ούτω ώστε τα γαλλικά και τα γερμανικά να ξεπεράσουν τα ισπανικά, τα οποία δεν μιλούνται μόνο στην Ευρώπη, αλλά τα μιλάνε επιπλέον άλλα 700 εκατομμύρια ανά την Ιφίλιο. Πολύ περισσότεροι από ό,τι τους Ευρωπαίους και πολύ πιο μπροστά από τα Ιταλικά. Διότι τα Ιταλικά και τα Ισπανικά τα, τα αναγνωρίζαμε στο γραφείο σήμανσης ως επίσημες γλώσσες. Nokia, Philips, Blackberry, Siemens κλπ. χρησιμοποιούν αυτές τις δύο γλώσσες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για μια ηλίθια διαδικασία τροχοπέδησης από μια μικροπροϊσταμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε Ας χρησιμοποιήσουμε εμείς ε, την ενισχυμένη συνεργασία. Ενισχυμένη συνεργασία η οποία μετά θα επιβαρύνει όλους τους υπόλοιπους. Διακόπτει ο πρόεδρος τον κύριο Μασίπ. Ευχαριστώ κύριε Μασίπ Ιδαλγό. Ο συνάδελφος Μέλτσερ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πολυγλωσία, όπως ξέρετε, είναι ένα αντικατόπισμα της ε, πολιτιστική και πολιτισμικής πολυμορφίας Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφωνία για τις γλώσσες μέσα στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ευρεσιτεχνίας, του διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ε, διαρκεί εδώ και 30 χρόνια. 30 χρόνια στα οποία οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ενδεχομένω ανταγωνιστικά μειονεκτήματα λόγω του υψηλού κόστους των μεταφράσεων. Είναι δύσκολο ίσως να καθορίσει κανένας αριθμητικά τι κοστίζει ε, η εικόνα μιας επιχειρήσης ε, και η πρόσβαση στην αγορά. Ίσως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ότι θα πρέπει να μεταβραστούν τώρα τα έγγραφα μόνο στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Αυτό θα διευκολύνει οπωσδήποτε το γραφειοκρατικό άχθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν εφαρμοστεί συνεπώς αυτό το καθεστώς των τριών γλώσσων, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, θα διευκολύνθει πολύ η κατάσταση. Και αυτό θα ενδυναμώσει επίσης και την ε, θέση της γερμανικής γλώσσας που από ό,τι είδαμε και το 2006 είναι η πιο πολύ ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Αλφο Μέρσερ. Περνάμε στη διαδικασία του ΚΑΣΤΙΑΗ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Υπουργέ, η δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα επιτρέψει την ε, τεχνολογική πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσουμε το θέμα του διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως για το κλασικό καθεστώς έχω αμφιβολίες. Κατά τη γνώμη μου ε, η καλύτερη λύση θα ήταν να εκδίδεται μόνο στα αγγλικά το δίπλωμα. Αν όμως είναι να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το θέμα γιατί είναι παγκόσμιο ανταγωνισμός ε, και το, ε, τα πορτογαλικά κατέχουν τρίτη θέση μετά τα αγγλικά και την Ισπανία ε, στον αριθμό των ομιλούντων αυτέ τι γλώσσε στον κόσμο. Ευχαριστώ, συνάδελφο Καρβάλιο. Σέρτσο που έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντα προτεραιότητα το θέμα της γνώσης Λυπήθηκα από όξα ότι η Βελική Προεδρία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την οδηγία για τι Ευρωπαϊκέ ευρυστεχνίες όσο έπρεπε και ελπίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει αυτό η Ουγγρική Προεδρία του επόμενου μήνε για να μπορέσει να προχωρήσει με την ενδυναμωμένη συνεργασία. Ο χρόνος είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξανακερδίσουμε. Χάνουμε χρόνο και δεν μπορούμε να το ξανακερδίσουμε κερδίσουμε. Χρειαζόμαστε να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις, χρειαζόμαστε να προωθήσουμε τις ευρυστεχνίες για την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα διπλώματα ευρυστεχνίας είτε με την κοινή ευρωπαϊκή ε, οδηγία είτε με την ε, ενδυναμωμένη συνεργασία να προχωρήσει. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους επιτυχία. Ουγγαρέζα και θα χάσουμε εμείς την Ουγγρική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι όλοι θα ωφεληθούν από το να μεταφράζονται στις τρεις γλώσσες τα βρεσιτεχνές. Ευχαριστώ κύριε Έρτσο. Ο κύριος Μάντες έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μπαρνιέ για την τόλμη που έδειξε να παρουσιάσει αυτά τα πράγματα εδώ γιατί στην ακρόση μας είχε υποσχεθεί να βρει τη λύση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας και θα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λένε για τις προσπαθίες. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε συμφωνούμε με την ενδυναμένη ε, συνεργασία ή όχι. Το πρώτο θέμα είναι αυτό που θα πρέπει να λύσουμε. Το δεύτερο θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε λιγάκι. Να κάνουμε δηλαδή μια διάκριση μεταξύ μιας γλώσσας σαν πολιτιστική έκφραση και γλώσσας για πρακτικούς λόγους. Στην πράξη όμως αυτό είναι σαφές, έχει αποδειχθεί καλό. Τώρα μπλοκάρουμε με την διαφωνία αυτή για τις γλώσσες την όλη πρόταση. Οι χώρες που δεν θέλουν να συνεργαστούν εδώ θα μπορέσουν να συνεργαστούν αργότερα. Ευχαριστώ στην Uh, Πρόεδρε, όταν πρωτοήρθα στο Κοινοβούλιο το 1999, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία ήταν στην εμμυρίσια διάταξη. Με τον Κλώσχα Χάινε Λένε συνεργαζόμασταν για την έκθεση τη κυρία Παλάσιο τότε και χάρηκα που σημειώνεται κάποια σοβαρή πρόοδο. Αρχίζει να σημειώνεται σοβαρή πρόοδο. Αλλά α μην υποτιμούμε, συνάδελφοι, τη σημασία αυτή τη πρόταση για την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Συζητούμε τώρα ένα εφάνταστο νέο σχέδιο περί ένωση τη καινοτομία. Αυτή η γυραιά ήπειρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφευρίσκει περισσότερα, να δημιουργούμε εφευρέσει και να τι εκμεταλλευόμαστε κιόλα. Είναι απολύτω απαραίτητο να έχουμε ανταγωνιστικό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Για, για αυτή την κίνηση τώρα, για την ενισχυμένη συνεργασία, ναι, είναι ε, ε, ένα τρίκ, αν θέλετε, για να προχωρήσει η διαδικασία επιτέλου. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να ρυθμίσουμε συνολικά το θέμα, διότι σε παγκόσμιο επίπεδο όλοι επιζητούν την Ένωση για την Καινοτομία. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και περαστικά σας, κύριε Χάρμαρ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η διαδικασία είναι αποκαλυπτική και από τη μορφή που έχει πάρει και από το περιεχόμενό τη. Δηλαδή, οι θύνοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν σε καθημερινή βάση να υπεραμείνονται των συμφερόντων του ε, παραβιάζοντα ε, τα κεκτημένα. Η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, με αυτή τη διαδικασία, τη ενισχυμένη διαδικασία, θα δημιουργήσει προβλήματα και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα για το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνία ε, θα έχει πάρα πολλέ επιπτώσει. Ε, Ποιο είναι ο στόχο να επιβάλλουμε ένα τέτοιο σύστημα και θα έχουν τα γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά ε, μια πλεονεκτική θέση. Τι θα γίνει με όλε οι υπόλοιπε γλώσσε. Γι' αυτό είπα αυτά που είπα στην αρχή τη παρέμβασή μου. Το, η Πορτογαλία έχει, τα πορτογαλικά συγγνώμη, έχουν την τρίτη θέση στον κόσμο ω προ τον αριθμό των ατόμων που ομιλούν αυτέ τι γλώσσε και είναι σημαντικό λοιπόν να το λαμβάνουμε υπόψη και για την καινοτομία θα πρέπει ναι με να κάνουμε τι κινήσει, αλλά όχι μέσα από αυτή τη επίθεση, δηλαδή τη βάζουν το πρόσχημα τη εξοικονόμηση του κόστου και έτσι προσπαθούν να περάσουν όλα του τα σχέδια. Ευχαριστούμε ε, κύριε Φερέιρο, ο συνάδελφο ε, Πάσκουα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Από το 2000 και μετά επιζητεί ε, καλύτερη συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ε, κατοχήρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. τεχνίας. Ε, σας παραπέμπω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ενστάσεις από πλευρά των κρατών μελών για το γλωσσικό καθεστώς και τις μεταφράσεις των διπλωμάτων ε, σε αντιπαραβολή με το ισχύον σύστημα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ληφθεί ε, απόφαση... κοινή απόφαση και να προχωρήσει η διαδικασία. Βέβαια, ταυτόχρονα κάποια κράτη-μέλη θέλουν να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα των εφευρετών σε παγκόσμιο επίπεδο και θέλουν να εκινήσουν αυτή τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία. Είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα θέσει κανένα φραγμό στην εκκίνηση αυτής της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για τα κράτη που το επιθυμούν. Σας ευχαριστούμε συνάδελφο Πάσκα. Ο συνάδελφος Σουάπ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά έλεγχαν, ακούστηκαν πολλά καλά επιχειρήματα. Θα ανακεφαλαιώσω λίγο. Καταρχήν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε οπωσδήποτε και να υποστηρίξουμε την πρόταση του συναδέλφου Λένε και να δεχτούμε την πρόταση του, του Επιτρόπου Μπαρνιέρ. Και ε, θα ήθελα εδώ πραγματικά να αναφέρουμε την πολύ επιτυχή εργασία της Βελγικής ε, Προεδρίας που ήταν επιτυχής και σε άλλους τομείς. Καταρχήν εδώ πρόκειται για μια απόφαση διαδικασίας. Δεν τέτοιο το θέμα ποιε θα είναι οι γλώσσες στην Ευρώπη που μιλούν από πόσους ανθρώπους και ποια είναι η πιο ωραία, αλλά πρόκειται για μια απόφαση που θα επιτρέψουμε στο Συμβούλιο να πάρει. Η συνάδελφο των Πρασίνων που μίλησε προηγουμένω έχει δίκιο ότι αυτή την απόφαση θα πρέπει να την εξετάσουμε προσεκτικά. Αλλά δεν πρόκειται για την επιτυχία μιας υποομάδας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θέλει να ακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς γλωσσικό. 25 από τις 27 χώρες θέλουν να ακολουθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσεκτικά μπορούμε να υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τώρα ευχαριστώ. Συνάδελφος Γκίρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας πρέπει να ενισχύσει την καινοτομία. Αυτός είναι ο στόχος του και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε ποια θα είναι η ιδανική μορφή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπάρχουν μακρές, μακρά διπλώματα, σύντομα. Θα πρέπει τα μακρύτερα να είναι πιο καλά από τα πιο σύντομα ίσως. και θα πρέπει γι' αυτό να φερθούμε σαν Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, υποστήριζα το ευρωπαϊκό το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή ε, καινοτομία και θα μπορέσουμε έτσι να προφυλαχθούμε και από τις ε, ε απομιμήσεις. μετά από 10 χρόνια το Συμβούλιο μόλις έφτασε στην δυνατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας. Ε, χαίρομαι που η τσεχική δημοκρασία ξανασκέφτηκε τη θέση της. Είναι πάρα πολύ λεπτά το θέμα όταν εξετάζεται η ενδυναμωμένη συνεργασία. Αυτό συνήθω λέγεται ότι είναι ένα θέμα που αφορά τι μεγάλε χώρε. αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι προ όφελο όλων των εφευρετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο στην τσεχική γλώσσα, θα είναι καλό να έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρυστεχνία και ελπίζω το Συμβούλιο θα μπορέσει να προωθήσει τα πράγματα πολύ καλύτερα. Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις ευρωπαϊκές ε, ευρεσιτεχνίες. Η κυρία Βάσλικ, για να ολοκληρώνουμε. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πάρα πολλά σχόλια σήμερα σχετικά με την ανάγκη κατοχήρασης ε, των εφευρέσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίες. Ε, οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται ένα αποτελεσματικό σύστημα για να είναι ανταγωνιστικές ε, σε σχέση με πολύ καινοτόμες επιχειρήσεις από τις αναδυόμενες οικονομίες. Ας μην λησμονούμε όμως ότι η διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας δεν είναι η πλέον επωφελής και δεν εξυπηρετεί υπηρετεί το στόχο του, της ενιαίας αγοράς. Εγώ είμαι θειασότης ε, της ενιαίας ε, εσωτερικής αγοράς, ε, οπότε δεν θα ταχθώ υπέρ αυτού του συστήματος και απευθύνω έκκληση προς όλους όσους εμπλέκονται ε, στην εξέταση του ζητήματος ε, για να πραγματευτούν λύσεις ε, για όλους. Εδώ αναφέρουν προφανώς το γλωσσικό καθεστώς. Υπάρχουν κάποιοι που δεν κατανοούν ούτε γαλλικά, ούτε αγγλικά, ούτε γερμανικά. νομίζω ότι είναι πλήμελες να βασίσουμε ολόκληρο το σύστημα σε μία μόνα γλώσσα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Χάνσλικ. Ολοκληρώσαμε το κάτσο τώρα και το λόγο θα έχει ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Εγώ θα σταθώ στην τελευταία σας φράση για να σταθούμε λίγο στην ουσία πέρα από τη διαδικασία. Είπαμε ότι έχουμε εργαστεί σκληρά υπό Βελγική Προεδρία και εδώ και μερικές εβδομάδες υπό Ουγγρική. Αν μια επιχείρηση βουλγαρική, σλοβακική, λετωνική, πορτογαλική θέλει να ζητήσει την ευρυσιτεχνία στη γλώσσα της μπορεί να το κάνει και το κόστος της μετάφρασης θα επιστραφεί. Σε περίπτωση διαφωνίας η επιχείρηση θα λάβει μία μετάφραση στη γλώσσα της. Αν δεν σεβαστεί την ευρυσιτεχνία προηγουμένως γιατί δεν έχει καταλάβει τη μετάφραση, τότε θα αποζημιωθεί. Εγώ πρότεινα μια επιχείρηση που θέλει να καταθέσει μια ευρυσιτεχνία να, να μπορεί να την καταθέσει και στη γλώσσα της. Η νομική προστασία θα διασφαλίζεται σε μια από τις τρεις γλώσσες που βασίζεται στις τρεις βασικές γλώσσες της Σύμβασης για τις Ευρυσιτεχνίες. με τη Βελγική Προεδρία προσθέσαμε μία πρόταση που θα τη συζητήσουμε. Ότι δηλαδή πέρα από τις τρεις γλώσσες της νομικής προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες δύο γλώσσες χωρίς μετάφραση του εγχειριδίου ας πούμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αγγλικά, θέλουμε τα αγγλικά, τα πορτογαλικά, τα λετονικά ή τα ολλανδικά και αυτή η μετάφραση επίσης θα είναι δωρεάν. Μία από τις τρεις γλώσσες για τη νομική προστασία και άλλες δύο για την ενημέρωση και πληροφόρηση. Δεν θα υπάρχουν διακρίσεις. Λοιπόν, ακόμη και για τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες που δεν έχουν δεχθεί την ενισχυμένη συνεργασία. Αν μία η ισπανική επιχείρηση θέλει να πάρει εύρηση τεχνία μπορεί να το κάνει άσχετα αν η Ισπανία συμμετέχει ή όχι. Περί περί αυτού πρόκειται. Εγώ εργάστηκα σκληρά, χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, χωρίς να λαμβάνω θέση για τον έναν και για τον άλλον. Στόχος ήταν να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πρόταση η οποία είναι πολιτικά αποδεκτή από τις 25 χώρες και για τις επιχειρήσεις των 27 χωρών μελών. Η κυρία Χέρτζοκ τόνισε πολύ σωστά την, όπως και ο κύριος Βάπεξ άλλου, την σημασία όλης αυτής της ιστορίας σε οικονομικό επίπεδο. Εμείς πρέπει να ενθαρρύνουμε, να προστατεύσουμε να χρηματοδοτήσουμε, να αποζημιώσουμε την καινοτομία. Να την ενισχύσουμε, να την προστατεύσουμε λοιπόν. Και αυτό αφορά σε πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα λόγω της έλλειψης ευρωπαϊκού, ε, ευρωπαϊκής ευρυσιτεχνίας δεν έχουν την δυνατότητα να προστατεύσουν την ευρυσιτεχνία τους. Και αν εμείς δεν προστατεύουμε την ευρυσοτεχνία, αυτό που είπε η κυρία Ροήτοβα για τις μαϊμούδες, οι οποίες είναι καρπός της έλλειψης προστασίας της Και όταν μπουν τα προϊόντα μαϊμούδες στην εσωτερική αγορά, καταστρέφουν την απασχόληση, την ασφάλεια, ακόμη και την δημόσια υγεία. Σκεφτείτε εσείς ε, φάρμακα. Είναι πολύ σοβαρά λοιπόν όλα αυτά. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, να βρούμε μια λογική λύση, μια αποδεκτή λύση. Να απαντήσω τώρα του κυρίου, Μασίπη, του κυρίου Τουρίλ για την ενισχυμένη συνεργασία που συσπηρώνει 25 χώρες των 27 και που χρησιμοποιείται για τον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο γιατί βρισκόμαστε σε μια εντελώς εξωτερική κατάσταση στην περίπτωση δηλαδή της ενιαίας αγοράς όπου χρειάζεται ομοφωνία. Για, ό, για όλους τις υπόλοιπους κανονισμούς ε, χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία και εδώ στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόμαστε ομοφωνία. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας κίνδυνος κατακαιρματισμού και η Κομισιόν περιφρουρεί για να το αποφύγει. Ευχαριστώ τον κύριο Λένε για τον βολονταρισμό του και τη στράτευσή του και ευχαριστώ και όλο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Επίτροπε κύριε Μπαρνιέ. Στον όνομα του Συμβουλίου κύριε Γκέωρη έχει το λόγο τώρα ma este az első felszólalásomban beszéltem már egy olyan nyelven amelyik az európai szabadalom. Στην πρώτη μου ομιλία θα χρησιμοποιώ μια γλώσσα που θα είναι, χρησιμοποίησα μια γλώσσα που είναι μια από τις ε, γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου, αλλά τώρα θα μιλήσω την ε, μητρική μου η οποία δεν προβλέπεται στο νέο γλωσσικό καθεστώς. Απευθύνομαι κυρίως στους Ισπανούς και Ιταλούς συναδέλφους στην ε, αίθουσα. Ε, πιστέψτε μας ότι ε, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο γλωσσικό καθεστώς και στην προστασία των μικρότερων γλωσσών. εκπροσωπούσα ένα κράτος μέχρι πριν από έξι εβδομάδες ε, στο κοινοβούλιο και η χώρα αυτή είχε διαφορετική θέση σε σχέση ε, με το ζήτημα, το γλωσσικό καθεστώς. Η Ουγγρική κυβέρνηση του τελευταίους μήνες έχει αλλάξει τη στάση της. Ε, δεν ήταν εύκολο να ληφθεί αυτή η απόφαση και ποιο ήταν το σημείο καμπής λοιπόν ώστε να ληφθεί η απόφαση από την Ουγγρική κυβέρνηση. Συμμετείχαμε σε εντατικέ διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και μας παρακάλεσαν να τροποποιήσουμε τη θέση μας, να μην ε, παρεμποδίσουμε την υιοθέτηση ενός ενιαίου διπλωμάτος ευρεσιτεχνίας, ε, γιατί ε, αν συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα θα εξυποκονομήσουν υψηλά ποσά για την προστασία των εφευρέσεών τους. Τώρα, η κατάσταση πώς έχει. 25 κράτη-μέλη συμφωνούν και δύο διαφωνούν. Δεν είναι ιδανική η κατάσταση, κυρίως όταν ε, ε, επιθυμούμε να οικοδομήσουμε μία ενιαία αγορά. Πάντως ευελπιστούμε ότι θα τονωθεί η ανάπτυξη με το νέο σύστημα, κυρίως όπως είπαν σωστά και οι συνάδελφοι, ε, την ώρα που προσπαθούμε να εξέλθουμε από την οικονομική κρίση. Ποιο είναι ο ακρογωνίος λίθος ενός νέου ανταγωνιστικού συστήματος είναι ακριβώς το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Όπως τόνισε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ, ε, θεωρώ και εγώ ότι όλες οι ισπανικές και οι ιταλικές επιχειρήσεις θα υποφεληθούν από το νέο σύστημα εάν πραγματοθεί στο μέλλον. Θα ήθελα να προσθέσω και δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, μας ρώτησε κάποιος... Ε, προς τι σπουδή, ε, γιατί ε, έχετε επισπεύσει τη διαδικασία εφόσον τον Ιούνιο υπέβαλε την έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Αξιότιμοι Βουλευτές. Νομίζω ότι απαντήσατε από μόνοι σας την ερώτηση. Ακούσαμε ότι εδώ και 10 χρόνια είναι υποσυζήτηση το γλωσσικό καθεστώς, οπότε δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για σπουδή. Ε, δεύτερον, ε, ε, μπορούμε να αναρωτηθούμε, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια γενικώ αποδεκτή λύση, αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, η Βελγική Προεδρία κατέβαλε πραγματικά κάθε δυνατή προσπάθεια. Δείτε όλες τις προτάσεις που εξετάστηκαν, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση και ευελπιστώντας ότι θα γινόταν αποδεκτή από τα 27 κράτη-μέλη δυστυχώς, τον ε, Δεκέμβριο 12 κράτη-μέλη ζήτησαν ενισχυμένη συνεργασία επειδή δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε συνενετική λύση. για αυξηθεί ο αριθμός. Σας είπα ότι 25 τώρα κράτη-μέλη συμφωνούν. Η Προεδρία δεν είχε άλλη επιλογή. Όφιλε να επιλέξει τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία και γι' αυτό ζητώ την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην ε, ψηφοφορία. Ε, σκεφτείτε την ενιαία εσωτερική αγορά. θα πρέπει να την τονώσουμε βάσει μελετών που έχουν γίνει προκύπτει ότι μία από τις τροχοπέδες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστορικής αγοράς είναι ακριβώς η έλλειψη του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κυρίως αληθεύει αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύσκολα μπορούν να ε, γίνουν πιο ανταγωνιστικές αν δεν υπάρχει αυτό το δίπλωμα. Ευχαριστώ κυρία Γιώργη. Για να ολοκληρώσουμε ο συγητής κύριος Λένα. Εξότιμες κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, τρεις παρατηρήσεις τελικά. Ο οποίος Παρνιέ ήδη είπε ότι η ενισχυμένη δημοκρασία, ε, συνεργασία έχει ακριβώς στον στόχο να ξεπεράσει τα προβλήματα με την ε, ομοφωνία. Η ομοφωνία είναι η εξαίρεση συνθήκης της αγώνας. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις και αυτό είναι ο στόχος της ε, ε, ενισχυμένης συνεργασίας. Τρεις γλώσσες. Μα αυτό δεν είναι το εξτάζουμε σήμερα, εξτάζουμε μόνο τη διαδικασία. Θα ήθελα να σας πω το εξή. Και στην έκθεση Παλάσσου είχαμε συζητήσει τότε ότι ακόμη πιο οικονομική θα ήταν η μία γλώσσα αλλά αναφέρθηκε επίσης ότι εδώ έχουμε και μια συμφωνία του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που εργάζονται πάνω στις γλώσσες που έχουν συμφωνηθεί. Μια ε, αλλαγή του συστήματος θα σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάχθει όλη η συμφωνία για τις... Ε, ευρωπαϊκές για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρυσυχνίας και αν αλλάξουμε αυτό το καθεστώ, θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τι 27 χώρες, θα, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τι 39 χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα έτσι, που θα το συζητήσουμε όταν συζητήσουμε την πρόταση τη Κομισιόν Επιτουσίας και οι νομικέ υπηρεσίε και των τριών θεσμικών οργάνων ήταν υπέρ τη ενισχυμένη συνεργασία. Τέλο, οι άνθρωποι τη πράξη δεν καταλαβαίνουν την πολιτική συζήτηση που κάνουμε εδώ και από σκοπιά εκείνων των ανθρώπων εκείνο που δινώνουν δηλαδή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εργάζονται έτσι και αλλιώς σε μία γλώσσα. Δηλαδή αυτή η συζήτηση για τη γλώσσα είναι κάτι που οι άμεσα διαφορόμενοι δεν καταλαβαίνουν καθόλου. Μετά, όσον αφορά το θέμα των διακρίσεων, εάν κατάλαβα καλά και είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα σωστά, αυτή η νέα ευρωπαϊκή ε, δίπλωμα ευρυστεχνίας είναι κάτι που είναι ανοιχτό για όλους τους ευευρέτες, όχι μόνο εκείνους που ανήκουν σε χώρες που έχουν συμφωνήσει, σε όλους τους ευευρέτες όλου του κόσμου θα έλεγα. Δεν υπάρχει κανένα μονέκτημα για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην ε, ε, ενισχυμένη στην εργασία. Δηλαδή, αν θέλω να επιβάλλω σε κάποιε από αυτές τις χώρες μια ευρυζεχνία, θα πρέπει να μεταφράσω τους άλλου. Λοιπόν, και εν καταλήξει, κανένα δεν θα εμποδιστεί αν θέλει να μεταφράσει τις, ε, τα διπλώματα αυτά ευρυζεχνίες σε όλε τι γλώσσε. Αν κάποια χώρα θεωρεί ότι είναι σωστό να μεταφραστούν τα διπλώματα αυτά ευρεστιχνία στη γλώσσα του, ας το κάνει, αλλά όχι εις βάρος των εφευρετών. Όχι, εκείνος που έχει ε, απαιτήσει πρέπει να είναι υπεύθυνο. Όποιο καλέσει τα όργανα θα τα πληρώσει κιόλα. Λοιπόν, εάν κάποιο θεωρεί ότι η γλώσσα του είναι τόσο σημαντική που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα διπλώματα βρυσαγνία Ευρώπη, α το κάνει. και ας το πληρώσει και μόνος του. Τελευταία ήταν αυτή η παρατήρηση που είχα να κάνω για να ξέρουμε τι συζητάμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ συνάδελφο. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση. Η ψηφορία θα γίνει αύριο. Επανώση με τη ημερησία διάταξη. Έκθεση Μπελέτ. Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα να ραδινέ στα τρόφιμα και ζωοτροφικά.